Ψηφίζουμε. Ψηφοφορία επί της εκθέσεως του κυρίου Μπέγκε. Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας. Θα έχουμε ονομαστική ψηφοφορία για την έκθεση αυτή. Χρειαζόμαστε ειδική πλειοψηφία. Άρχεται η ψηφοφορία. Wszyscy głosowali. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. 544 ψήφοι υπέρ, 18 κατά 14 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Τώρα. Θα ψηφίσουμε τώρα την έκθεση πάλι για το δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013 με ονομαστική ψηφοφορία πάλι έκθεση του κυρίου Μπέγκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. 536 ψήφοι υπέρ 18 κατά 22 αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε σχέδιο τροπολογιών στο Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το οικονομικό έτος 2010. Κύριο Σουριανή είναι Θα ήθελε το λόγο ο εισηγητή, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Είμαστε ενώπιον της ε, πιο σύντομη ψηφοφορία, αν θέλετε, στα θέματα προπολογισμού στα πλαίσια τη συνθήκη τη Νίκαια. Και είναι και τελευταία ψηφοφορία στα πλαίσια τη ε, συνθήκη αυτή. Πώ είναι δυνατόν να είναι τόσο σύντομο ο κατάλογο ε, των ψηφοφοριών, χάρη στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των ομάδων. Ω εισηγητή, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλε τι ομάδε οι οποίε συνέβαλαν στην προετοιμασία τη ψηφοφορία αυτή. Και επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη γραμματεία για το έργο της. Χωρίς αυτήν θα ήταν εξίσου αδύνατο να βρεθούμε σήμερα εδώ με δύο μόνο σελίδες. Σας ευχαριστώ όλους σας και νομίζω ότι ο σύντομος αυτός κατάλογος ψηφοφοριών Πρόεδρος Διακόπτη Λοιπόν, ψηφίζουμε τη δέσμη παριθμών 1, παρακαλώ. Υπέρ κατά αποχές δεκτό προχωρούμε τροπολογία 48 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές θα γίνει έλεγχος χρειάζεται ειδική πλειοψηφία άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας της ψηφοφορίας «342 υπέρ 219 κατά τρεις αποχές δεν εγκρίνεται γιατί δεν επιτεύχθηκε η ειδική πλειοψηφία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 382. Σε τμήματα, δύο τμήματα συγκεκριμένα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα, θα γίνει με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Ε, ψήφισαν υπέρ 476, 80 κατά 12 αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την δεύτερη ομάδα των υπολογιών υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται η ομάδα. Ψηφίζουμε την τρίτη ομάδα τροπολογιών υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τέταρτη ομάδα τροπολογιών υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Πέμπτη ομάδα τροπολογιών υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έκτη ομάδα των απολογιών υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έβδομη ομάδα των απολογιών υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 290 κατά τμήματα. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Κατά διορθώνει ο Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος για την επαλήθευση της, του δεύτερου τμήματος. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Εψήφισαν υπέρ 415, 151 κατά 4 αποχές. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. τμήμα τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται το τρίτο τμήμα. Επί του κανονισμού. Έτοιμα. Κύριε Πρόεδρε, προτείνω για την ομάδα των άλλων θεσμικών οργάνων να ψηφίσουμε ομού. Δεν περιμένω να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Κοιτάξτε, η κατάσταση έχει ως εξής. Ψηφίζουμε επί του προπολογισμού των διαφόρων οργάνων βάσει των αρχών και βάσει των αρχών των υποχρεώσεών μας πρέπει να ψηφίσουμε ξεχωριστά για κάθε όργανο. Όχι ενιαία γιατί αυτό είναι αντίθετο με τον κανονισμό και τη διαδικασία που μέχρι τώρα ακολουθήσαμε. Δικαστήριο. Ομάδα τοπολογιών 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ελεγκτικό συνέδριο. Ομάδα 9 τοπολογιών υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, δέκατη ομάδα των υπολογιών, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επιτροπή Περιφερειών, ενδέκατη ομάδα των υπολογιών, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ομάδα 12, υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου Προστασίας Δεδομένων. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ωραία. Έτσι, κλείσαμε το τμήμα αυτό. Δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, το Συμβούλιο σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε πλέον τη συμφωνία την οποία ε, επιτέχθησε τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτου μαζί με το αποτέλεσμα της δεύτερης ανάγνωσης ε, στο Συμβούλιο βλέπουμε ότι η δεύτερη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο πλέον παρήγαγε ένα κοινό κείμενο σύμφωνα με την 314 ε, το άρθρο 314 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Αποδεχόμαστε το κείμενο αυτό και χαιρόμαστε που η Προεδρία μπορεί πλέον να δηλώσει ότι είναι πλέον εγκεκριμένος ο προπολογισμό. Θα ήθελα να σημειώσω ότι από τη στιγμή που θα εγκριθεί ο προπολογισμό θα πρέπει να υπογραφεί και από τα δύο μέρη σύμφωνα με την σχετική νομική πράξη, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει σχετική διάταξη περί ισότητας των δύο μερών. Αυτό δεν έχει ληφθεί υπόψη ωστόσο δεν ε, προβάλλουμε οποιαδήποτε ένσταση σε αυτά που έχουν συμφωνηθεί. Ελπίζουμε ότι του χρόνου στην διαδικασία έγκριση του προπολογισμού θα υπάρξει χρόνο να διευκρινιστεί το θέμα. Θα ήθελα επίση επί του παρόντο να διευκρινίσω ότι θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σούργιαν, τον κύριο Μάνκα για την επικοδομητική του στάση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η οποία και πάλι αποτυπώνεται στην εξαιρετική συνεργασία, την οποία πραγματικά μπορώ να πω ότι απολαύσαμε. Και τέλος ένα προσωπικό σχόλιο, επιτρέψτε μου, ως ε, μέλος της Προεδρίας. Πρέπει να πω ότι είναι μία από τις καλύτερες θέσεις που έχω περάσει ποτέ στην καριέρα μου και ήταν μεγάλη μου τιμή να γνωρίσω την Ευρώπη υπό την ε, άποψη αυτή και ήταν ε, να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ. Κλείσαμε το τμήμα αυτό της ψηφοφορίας. Θέλω και εγώ προσωπικά να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή μας κύριο Σουριάν και τον κύριο Μάντα καθώς και τον κύριο Μπέγκε βέβαια και ευχαριστώ και όλους όσοι ασχολήθηκαν με τον προϋπολογισμό δύσκολο προϋπολογισμό μπράβο λοιπόν και μπράβο και στο κοινοβούλιο γιατί πήραμε γρήγορα και μαζί την απόφαση κάνετε πολύ καλή δουλειά συνάδελφοι συγχαρητήρια ε, muszę Państwu odczytać bardzo ważne punkty να σας διαβάσω τώρα ένα σημαντικό κείμενο που αφορά την έκτακτη διαδικασία έγκρισης του προπολογισμού. Είναι πολύ σημαντικό. Περάσαμε από τη συνθήκη της Νίκης στη συνθήκη της Λισαβόνας. Ένα δύσκολο πέρασμα. Ξεκινήσαμε με τη Νίκαια, κλείνουμε με τη Λισαβόνα. Η δήλωση αυτή είναι αναγκαία και παρακαλώ να ακούσετε. Η διαδικασία προπολογισμού για το έτος 2010 ήταν εξαιρετική. Ξεκίνησε βάσει το άρθρο 272 της ε, Συνθήκης Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η τελευταία φάση της διαδικασίας αυτής, ωστόσο, ολοκληρώθηκε κάτω με ενισχύ τη συνθήκη της Λισαβόνας. Στις 18 Νοεμβρίου του 2009, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή αποφάσισαν να συνεχίσουν την ε, δημοσιονομική διαδικασία βάσει της συνθήκης ΕΟΚ, της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Κοινότητας και συμφώνησαν σε ό,τι αφορά την έκβαση τη δημοσιονομική διαδικασία, συμπεριλαμβάνοντα και την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο που μόλι τώρα έλαβε, με πλήρη σεβασμό των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου επιβεβαίωσε την συμφωνία στο Συμβούλιο σε σχέση με τον προπολογισμό που μόλι ψηφίσαμε. Τούτο σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πέτυχαν μια συμφωνία επί ενό κειμένου, τηρώντα του στόχου και τον σκοπό του άρθρου 314 της Συνθήκης λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία προπολογισμού που ξεκίνησε λοιπόν με βάση το άρθρο 272 της Συνθήκης που ιδρύει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και συνεχίστηκε με την ε, βάση του άρθρου 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκληρώθηκε βάσει του τελευταίου αυτού άρθρου, το άρθρο 314 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα στις, ε, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών πολιετών ε, του δημοσιονομικού ε, οικονομικού πλαισίου. Ο υπολογισμό κατά συνέπεια έχει ολοκληρωθεί και έχει εγκριθεί. Πρόκειται για μια σημαντική δήλωση. Η δήλωση αυτή Το πρόβλημα αυτό δεν θα το έχουμε από του χρόνου, διότι θα ισχύει πλέον μόνο η συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα, υπογράφω επίσημα το κείμενο αυτό. Να προσθέσω και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε. Ο κύριο Λαμασούρ, πρόεδρο τη Επιτροπή Προπολογισμών, έπαιξε και αυτό πολύ σημαντικό ρόλο. Θέλω λοιπόν να αναφέρω και το δικό του όνομα. Πρόκειται για ένα άτομο που συνεργάστηκε πραγματικά ενεργά και δραστήρια στην επίτευξη του στόχου μα. Στη, στο θεωρείο έχουμε μια αντιπροσωπεία από την Σερβία που καλωσορίζουμε. Σηκωθείτε αν θέλετε για να σας δούμε. Ε, proszę Państwa, jeszcze Μισό λεπτό ακόμα, συνάδελφοι, για τον προπολογισμό πάντα πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεση Σουριάν και Μάνκα για το σχέδιο Γενικού Προπολογισμού της Ευρωπαϊκής